Liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε και ίσως πρώτα απ' όλα μπορούμε να δούμε όλοι μαζί το βίντεο που θα προβληθεί. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μένα εκπροσωπώντας ε, τον Ραΐφ Μπαντάμπη να απευθυνθώ σε εσά. Ο κύριος Μπαντάουι σήμερα δεν μπορεί να είναι κοντά μας γιατί ε, ξέφρασε ελεύθερα την ε, άποψή του και κάλεσε και όλους τους υπόλοιπους να πράξουν το ίδιο. Για το λόγο αυτό ε, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση και χίλιους ραβδισμούς. Όταν ενημερωθήκαμε για το τραγικό γεγονός ότι ού μόνον αυτό αλλά επιπρόσθετα βρίσκεται και σε απομόνωση στη φυλακή γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί για να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ και γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά ε, να απευθυντώ σε εσά ε, στη σύζυγό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να την καλωσορίσω. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας ε, πολλούς ε, προσκεκλημένους ε, οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν και αυτοί στην απονομή του βραβείου του βραβείου Ζαχάροφ 2015. Έχουμε πολλούς εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος. Μεταξύ όμως αυτών υπάρχουν δύο προσκεκλημένοι, τους οποίους επιθυμώ ιδιαίτερα να καλωσορίσω. το έχω συμφωνήσει και με την κυρία Χαϊντά ότι θα απευθυνθώ ιδιαίτερα στην Όλκα Σόρεβα από το Ίδρυμα Πόρης Νέτσοφ και στη Μαρία Αλεχάνδρα Αρίστη Γκουίντα, εκπρόσωπο της ε, αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Αυτοί οι δύο εκπρόσωποι και αυτές οι δύο ομάδες ε, ήταν επίσης υποψήφοι για το βραβείο Ζαχάρου. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά εδώ κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου Ζαχάρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι που ήρθατε κοντά μας. Μέσω ημών, κυρία Χάιντα, θα θέλαμε να εξάρουμε και να τιμήσουμε τον θαραλέο αγώνα του συζύγου σας. Αξιότιμη κυρία Χάιντα, επιθυμώ να απευθυνθώ σε εσά προσωπικά, στην οικογένειά σας, στα παιδιά σας, στους φίλους σας και επιτρέψτε μου να τονίσω το θάρρος σας και την αποφασιστικότητά σας στον αγώνα που διεξάγεται για να έρθει πίσω ο σύζυγός σας στο σπίτι του. Δύο μικρά παιδιά, 12 και 8 ετών. Αυτά τα μικρά παιδιά περιμένουν την επιστροφή του πατέρα τους. Και επιτρέψτε μου να υποκληθούμε σε εσά και εσείς, ακριβώς επειδή αντιμετωπίσετε την θανατική ποινή, αναγκαστήκατε να φύγετε στον Καναδά, εκεί σας χορηγήθηκε άσυλο και από τον Καναδά ορμόμενοι αγωνίζεστε άοκνα και ακούραστα για την απελευθέρωση του συζύγου σας. Εκείνος και η φωνή του είναι απολύτως απαραίτητες, γι' αυτό λοιπόν εξ όλων μας απαιτώ εδώ εξ αυτού του βήματος και καλό τον ε, την εξοχότητα του βασιλιά Σαλμάν να δώσει χάρη στον ε, Μπαντάουι, στον κύριο Μπαντάουι και να επιτρέψει να επιστρέψει στην ε, οικογένειά του χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση. Παρά λοιπόν τους πολλούς κινδύνους, ο Μπαντάουι προσπαθεί πολύ ταραλέα μέσω των blog να προάγει την ελεύθερη σκέψη. Όταν λοιπόν το δικαίωμά του για την ελεύθερη έκφραση άποψης αμφισβητήθηκε, δεν δίστασε με τον blog του, κάλυψε ένα κενό, ένα κενό σε μία χώρα που το κενό αυτό είναι μία χένουσα πληγή γιατί δεν υπάρχει ελευθερία σκέψης και ελευθερία τύπου. Ήψωσε λοιπόν τη φωνή του για το ότι οι άνθρωποι δικαιούνται να λένε και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Απαιτεί λοιπόν να υπάρχει μια ανοιχτή κοινωνία, ανοιχτή και για τις απόψεις των υπολείπων. Όταν ήταν στη φυλακή, ε, μέσα από το τηλέφωνο ε, υπαγόρευσε αυτά που έπρεπε να αναφέρονται στο προήμιο του βιβλίου του. Λέει λοιπόν ότι τα τείχη της άγνοιας πρέπει να κατεδαφιστούν. Ο κύριος Μπαντάου ακολουθεί το στόχο που είναι ότι το πνευματικό έργο και οι διανοούμενοι είναι στο αλόβητο και δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός για την ελευθερία της σκέψης, εγγυήσει για την ελευθερία αυτή, σεβασμός των δικαιωμάτων των γυναικών, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τήρηση των βασικών δικαιωμάτων κάθε μεμονωμένου πολίτη και ατόμου. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο Ρεφ Μπαντάουι το 2006 συνέστησε το φόρουμ, το blog το δικό του ε, και ήταν απολύτως απαραίτητο, όπως επισήμανε, να υπάρξουν μεταρρύθμιση πολιτικό και θρησκευτικό επίπεδο. Θέλησε μέσω του blog του να προβάλλει αυτές τις απόψεις. Ε, η κυβέρνηση ε, αποφάσισε να κλείσει αυτό το φόρουμ η φιλελεύθεροι της ε, Σαουδικής Αραβίας. Του αντίον αυτός επανήλθε όμως με ένα νέο ιστότοπο, στον οποίο ιστότοπο έχουν κλικάρει χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι συζητούν για την πολιτική και για τη θρησκεία. Και όταν άρχισε να εμφανίζεται η Αραβική Άνοιξη, σε αυτό το δίκτυο και σε αυτή την πλατφόρμα υπήρχε μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Το κλείσιμο λοιπόν του ιστότοπου του κυρίου Μπαντάουι ήταν μια μεγάλη απώλεια για την ελευθερία της σκέψης στη χώρα του. Ο Μπαντάουι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όχι μόνο λογοκρίτηκε αλλά και συνελήφθη και ε, δέχτηκε τους πρώτους 50 ενώ το πλήτος επεφημούσε και αυτό σοκάρισε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους και κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή τη βιαιότητα. Λόγω λοιπόν της ε, κακής υγείας του Ραΐφ ε, ε, προσωρινά αναβλήθηκαν οι υπόλοιποι ραβδισμοί. Ο Ραΐφ Μπαντάου έγινε λοιπόν ένα σύμβολο, πηγή έμπνευση για όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται για τα θεμελιώδη δικαιώματα όχι μόνο στη δική του περιοχή αλλά και πολύ πέρα από αυτήν, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πράγματι λοιπόν ο Ραΐφ Μπαντάου σε αυτό τον αγώνα δεν είναι μόνος του. Ο δικηγόρος του, ο Μπαλέ Αλμπού Αλκαΐρα, 36 ετών και εκείνος εκτεί ε, ποινή κάθριξης 15 ετών ε, διότι ίδρυσε ε, και ένα παρατήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδικάστηκε και για τα tweet που είχε κυκλοφορήσει σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Δόκτωρ Νταρίν Καϊνταπόη ο οποίος επίσης ε, και αυτός ε, ίδρυσε ένα Ινστιτούτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτός είναι ο δέκατος που κλείστηκε στη φυλακή και αυτός καταδικάστηκε με ραβδισμούς και απαγόρευση εξόδου της χώρας για δέκα έτη. Πριν από λίγο καιρό ο Ρασάτ Παγιάτ, ένας ε, νέος ποιητής, καταδικάστηκε και αυτός για αποστασία, για αποκήρυξη της πίστης του. Και βεβαίω στη δική του την περίπτωση δεν υπήρχε δίκαιη δίκη, ούτε και ε, νομική εκπροσώπηση, κάτι το οποίο στυλίτευσε η παγκόσμια κοινότητα. Ο Αλ Μοχαμίτ Αλνίμιρ, 21 ετών, δεν ήταν ούτε καν 18 ετών όταν συνελήφθη γιατί και εκείνος ε, ε, συμμετείχε σε διαδηλώσεις στη Σαουδική Αραβία. Και γι' αυτό το λόγο και μόνο καταδικάστηκε σε θάνατο με σταύρωση. Είμαστε λοιπόν όχι μόνο ανήσυχοι, αλλά σοκαρισμένοι, σοκαρισμένοι για όλα αυτά ε, και για το ότι θα εκτελεστούν αυτές οι ποινές τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όπως το κάναμε λοιπόν για τον Ραϊφ Μπαντάουι, έτσι και στην περίπτωση των υπολείπων που σας ανέφερα, μέσω ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλούμε τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ε, να λάβουν υπόψη τους τα αιτήματά μας, να απελευθερώσουν τον Άλι Μοχάμετ Αλ να άρουν την, καταδική, ε, την θανατική καταδίκη, να μην εκτελεστεί αυτή η ποινή. Όμως αγαπητοί συνάδελφοι, οι περιπτώσεις αυτές είναι μόνο λίγες, κάποιες από πολλές περιπτώσεις οι οποίες ε, ακολουθούν και πολλούς άλλους ανθρώπους, οι οποίες ε, συνοδεύονται από θανατική ποινή. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τη Σαουδική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαουδικής Αραβίας, να πάυσει να επιβάλλει τέτοιου είδους ε, καταδίκες. Μα η χώρα έχει υπογράψει διεθνείς συνθήκες και επιτέλους να τη σεβαστεί. Η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει τη διεθνή συνθήκη καταδίκης βασανιστήριων για τα δικαιώματα επίσης των παιδιών, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση βάρος των γυναικών. Τα έχει υπογράψει όλα αυτά η Σαουδική Αραβία. Η διεθνής κοινότητα και η Σαουδική κοινότητα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήματα έναντι της κυβέρνησης ε, διότι η χώρα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει υπογραμμιστεί και προβληθεί επανειλημμένα ότι παρόλα αυτά στη χώρα όμως η οποία είναι μέλος των Εθνών δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα μια χώρα η οποία συμμετέχει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων ε, σε αυτή τη χώρα σε ένα και μόνο χρόνο εκτελέστηκαν 150 άνθρωποι η κοινωνία λοιπόν της Σαουδικής Αραβίας ε, ζητάει να υπάρχει επικοινωνία, να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως υπάρχουν έντονες λογοκριτικές τάσεις. 400 blog έχουν απαγορευτεί. Οι άνθρωποι λοιπόν που επιθυμούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους δέχονται βαρύτατες ποινές. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η διεθνή κοινότητα είμαστε ανοιχτοί για διάλογο. Διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σαουδική Αραβία. Αν αυτό στηριχτεί κοινοβουλευτικά μπορεί να συμβάλλει σε βελτίωση της κατάστασης, σε βελτίωση της αλληλοκατανόησης και τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Υπήρξαν βέβαια κάποιες ε, θετικές εξελίξεις, να το πούμε και αυτό. Ο Υπουργός ενέκρινε κάποιες ε, Κάποιου ιδιωτικού φορεί, Ελπίζουμε να μην μετατραπούν αυτοί σε κρατικού φορεί. Ε, αυτοί οι φορεί ε, υπάρχουν και έχουν μέλη από την ε, κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν και κάποια δικαιώματα των γυναικών τα οποία έχουν αναγνωριστεί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Εμεί αγωνιζόμεθα για τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Καμία διακριτική μεταχείριση. Καλούμε λοιπόν τη Σαουδική Αραβία να τηρήσει τι υποχρεώσει τη και να καταργήσει την ανδρική κατακυδαιμονία και κατακυδαιμόνευση των γυναικών, γιατί αυτό πια δεν έχει καμία σχέση με τον 21ο αιώνα. αξιότιμη κυρία Χάιντα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Καμία τρομοκρατία, αλλά και καμία θανατική ή οποιαδήποτε άλλη ποινή δεν θα μας εμποδίσουν να αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κανένα επιχείρημα περί ασφαλείας και κανένα λατρεμπόριο όπλων ή οποιαδήποτε μορφή εμπορίου όπλων δεν θα μας συγκρατήσει να προχωρήσουμε. Ο Ραΐφ Μπαντάουι είπε ταξί και παραθέτω. Η έκφραση της ελεύθερης άποψης είναι το οξυγόνο το χρειάζεται αυτό ο ε, λόγιος, ο διανοούμενος για να μπορέσει να εκφράσει τις απόψεις του. Τέλος της παράθεσης. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα το να δίναμε να απομείν, απονείμω το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2015 στο Ραΐφ Μπαντάουι. Και Θέλω να πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα μας δοθεί η δυνατότητα να τον καλωσορίσουμε εδώ τον ίδιο στην Ολομέλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την απονομή του βραβείου αυτού. Είναι τεράστια τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα πραγματικά ο σύζυγός μου να μπορεί ο ίδιος να παραλάβει το βραβείο αυτό. Θα ήθελα ωστόσο με την άδειά σας να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους τόσο στη Γαλλία όσο και αλλού. Ο σύζυγός μου επιθυμούσε ακριβώς αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να τηρήσουμε εδώ πέρα ενός λεπτού σιγή προς τιμή των θυμάτων. ألف شكر لكم ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Βρίσκομαι ενώπιόν σας Σας μιλάω με έναν τρόπο στεναρό σε εσά που είστε εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη να εκπροσωπώ το σύζυγό μου, ιδιαίτερα περήφανη που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα από τα πιο σημαντικά όργανα της δημοκρατίας παγκοσμίω. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενη σε ένα άρθρο που έχει γράψει ο σύζυγός μου. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ο καθαρός αέρας που αναπνέει κάθε στοχαστής. Είναι το καύσιμο που αναζωπυρώνει τη σκέψη του. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, τα έθνη και οι κοινωνίες κατάφεραν να προοδεύσουν χάρη στους στοχαστές τους. Χάρη στις ιδέες και χάρη στις φιλοσοφίες που τους προτείνονται, οι λαοί μπορούν να επιλέξουν το πλέον κατάλληλο σύστημα σκέψης και στη συνέχεια μπορούν να τον απτύξουν περαιτέρω προκειμένου να του οδηγήσει στην επιστήμη, στην πρόοδο, στον πολιτισμό και στην ευημερία. Η διεθνή κοινότητα και οι οργανώσει προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν από τα αραβικά καθεστώτα περισσότερε μεταρρυθμίσει στον τομέα τη ελευθερία τη έκφραση. Θεωρούν πω πρόκειται για ένα ουσιαστικό δικαίωμα. Είστε άνθρωπο, άρα έχετε το δικαίωμα να εκφράζεστε και να σκέφτεστε ελεύθερα και το δικαίωμα να εκφράζετε τη σκέψη σας. Έχετε το δικαίωμα να πιστεύετε και να στοχάζεστε, το δικαίωμα να αγαπάτε, να μισείτε, το δικαίωμα να είστε φιλελεύθερος ή Ισλαμιστής. Ωστόσο, οι Άραβες στοχαστές, ακόμα και όταν υποστηρίζουν η ελευθερία της σκέψης, συνηθίζουν να περιβάλλουν τις ιδέες τους με αρκετή ασάφεια, ώστε να γίνουν τα κείμενά τους αποδεκτά. Ιδίως όταν οι ελεύθερες και φωτισμένες σκέψεις τους θεωρούνται θρησκευτική αποστασία και βλασφημία. Καθώς για ορισμένες αραβικές κοινωνίες η ελεύθερη σκέψη αποτελεί διάλυση, θρησκευτική και ηθική παρέκκληση. Είναι φυσιολογική αυτή η κατάσταση, σας ρωτώ, προφανώς όχι. Δρούν αφύσικα και ο Άραβας, το χαστής και η κοινωνία. Ο στοχαστής οφείλει να εκφράζει τις ιδέες και την κοσμοθεωρία του με ειλικρίνεια και τόλμη, ακόμα και αν σφάλισε κάποια σημεία ή αν οι ιδέες του πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα της θρησκευτική παράδοσης. Η κοινωνία, από την άλλη, οφείλει να αγκαλιάσει όλες τις μορφές σκέψης και όλα τα πνευματικά κινήματα. Οφείλει η κοινωνία να αφουγκράζεται τις απόψεις των άλλων προκειμένου να μπορεί να τις κρίνει επικοδομητικά μέσω ενός δημιουργικού διαλόγου. Στόχος θα πρέπει να είναι να αξιολογούνται και να αναπτύσσονται περαιτέρω ιδέες και ένας εξωτερικός παρατηρητής θα έβλεπε ότι η αραβική κοινωνία αγκομαχά και στενάζει κάτω από τον ζυγό ενός θεοκρατικού καθεστώτος καθώς το μόνο που τη ζητείτε είναι να υποκλίνετε και να υποτάσετε τη στους κληρικούς. Κατά συνέπεια, οι κοινωνίες αυτές αναγκάζονται να αποταχθούν στον κλήρο με αποτέλεσμα όλες οι ε, φετφάδες και διάφορες θρησκευτικές ερμηνείες να καταλήγουν να θεωρούνται απόλυτες και ιερές αλήθειες. Κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι δέχονται πάρα πολλές απειλέ, μόνο και μόνο επειδή εκφράζονται ελεύθερα. Αυτό που φοβάμαι περισσότερα είναι μήπω ε, εξαιρετικοί Άραβες του πνεύματος εγκαταλείψουν τη χώρα αναζητώντας οξυγόνο μακριά από τον θρησκευτικό αυταρχισμό. Κυρίες και κύριοι, ο σύζυγό μου, προτού χρειαστεί να πάει στη φυλακή, είχε πει ότι η θρησκεία προσπαθεί πολλές φορές ε, να εκφοβήσει τους ανθρώπους ότι πολλέ φορέ οι κληρικοί φοβούνται ότι οι πνευματικοί άνθρωποι ενδεχομένω θα τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του. Ο Ραϊφ Μπαντάουι είναι ένα νέο Σαουδάραβα, ο οποίο βρίσκεται στην φυλακή ήδη από το 2012. Κατηγορήθηκε για θρησκευτική αποστασία. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση σε 300.000 δολάρια πρόστιμο και πρόκειται να λάβει χίλια, το παραλαμβάνω, χίλια χτυπήματα με μαστίγιο, τα οποία πρέπει να λάβει κάθε εβδομάδα 50 ραβδισμοί κάθε Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση της προσευχής. Επίσης, του απαγορεύεται να ταξιδέψει και να κάνει δηλώσεις στον τύπο και αυτό για μια περίοδο 10 ετών μετά την απελευθέρωσή του, αφού εκτίσει δηλαδή την ποινή του. Ο Ραΐφ δεν είναι εγκληματία, δεν είναι βιαστή. Ο Ραΐφ είναι ένα ελεύθερο στοχαστή, ένα ελεύθερο πνεύμα. Ποιο είναι το έγκλημα το οποίο διέπραξε. Πολύ απλά το ότι μίλησε ελεύθερα και ανοιχτά σε μια χώρα που δεν δέχεται άλλες απόψεις. Ο σύζυγός μου δεν είναι εγκληματίας. Δεν είναι διακινητής ναρκωτικών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δέχεται μια τόσο απάνθρωπη ποινή, μια τόσο σκληρή και ομή ποινή. Ο σύζυγό μου απλώ προσπάθησε να εκφράσει την άποψή του και να την καταγράψει στα γραπτά του. Ο σύζυγό μου ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο που θα μπορούσε να δεχθεί ελεύθερα τι απόψει όλων των ανθρώπων. Σε μια χώρα που θεοκρατείται, σε μια χώρα μονόχνοτη ενιαία σκέψη. Γι' αυτό το λόγο αποτελεί σήμερα σύμβολο τη ελευθερία όχι μόνο στην Σαουδική Αραβία αλλά παντού στον κόσμο. Ο Ραϊφ Μπαντάουι είναι πολύ απλά ένας ε, ειρηνικός ελεύθερος στοχαστής. Δεν ήθελε να ακολουθήσει το κοπάδι που τόσο τυφλά ακολουθεί τον κλήρο. Έναν κλήρο ο οποίος ζει σε μια άλλη εποχή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ένας κλήρος ο οποίος επιβάλλει ένα πολύ αυστηρό νόμο στη Σαουδική Αραβία. Όρθωσε λοιπόν το ανάστημά του, μίλησε, μίλησε ανοιχτά και αντιτάχθηκε στη βαρβαρότητα και στην ε, τυραννία. Και βλέπετε όμως ποια είναι η ποινή η οποία έλαβε. 50 πρώτες μαστιγώσεις οι οποίες οδήγησαν σε διεθνή κατακραυγή. Κατακραυγή που δεν έχει καπάσει ακόμα. Το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλέ χώρε, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Σε πάρα πολλέ χώρε υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνονται όρθιοι και λένε ελεύθερα Είμαι κι εγώ ο Ραϊφ Μπαντάουι. Το βραβείο λοιπόν αυτό που το απονέμεται σήμερα είναι θεωρώ ένα ιστορικό βραβείο και μια ιστορική στιγμή για τον αγώνα του καταδεικνύει πραγματικά το θάρρος σας, κύριε Πρόεδρε, το θάρρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το 15ο κατά σειρά βραβείο το οποίο λαμβάνει ο σύζυγός μου σε λιγότερο από ένα χρόνο. Σήμερα λοιπόν είναι ο πρώτος κατά σειρά πολίτη από την περιοχή του Περσικού κόλπου που λαμβάνει τόσα πολλά βραβεία και που λαμβάνει προφανώ και το βραβείο Ζαχάροφ. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πάρω το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και θα ήθελα να πω ότι ο, ο Ραΐφ Μπαντάουι είχε πει ότι όσοι θέλουν για μας το θάνατο, εμείς προασπίζουμε τη ζωή. Προασπίζουμε τη γνώση ενάντια στην άγνοια. Σας ευχαριστώ πολύ.

Νομίζω ότι δίναμε εξ ονόματος όλων για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τη σύζυγο του κυρίου Μπαντάουι. Είχα την δυνατότητα πριν από την ομιλία της να συζητήσω μαζί της μια μακρά συζήτηση και νομίζω ότι και εσείς θα αισθανθείτε όπως αισθάνθηκα και εγώ. Μου μίλησε για τα τρία της παιδιά ένα κοριτσάκι 12, ένα γόρι 11 και άλλο ένα κοριτσάκι 8 ετών. Αυτά τα τρία παιδιά περιμένουν στον Καναδά τον πατέρα τους. Η κυρία Χαϊντά μου είπε ότι ο κύριος Μπαντάουι κάθε φορά που τη μπαίνει στο τηλέφωνο ή που μιλάνε στο τηλέφωνο ε, της λέει ένα πράγμα «Πρόσεξε, μη με ξεχάσουν τα παιδιά». Και νομίζω όλοι μας ε, μπορούμε να αισθαντούμε τι σημαίνει αυτό για τον πατέρα αλλά και για τη μητέρα η οποία είναι αναγκασμένη να μιλάει κάτω από αυτές τις συνθήκες με το σύζυγό της και να ακούει αυτά που ακούει. Και του λέω κάθε φορά μη φοβάσαι, μη φοβάσαι Κανένας δεν θα σε ξεχάσει, δεν θα σε ξεχάσουν τα παιδιά μας και νομίζω ότι η σημερινή τελετή συνέβαλε στο να γνωρίζουν τα παιδιά ότι κανείς δεν θα ξεχάσει τον πατέρα τους. Αγωνιζόμαστε γι' αυτόν. Και κυρία Χαϊντά, θέλω να σας πω ότι όλοι οι παριστάμενοι στην αίθουσα σας θαυμάζουν για το θάρρος σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την εργασία μας που σύμφωνα με την, τον, κανό, τον κανόνα 252 και αφού διαβουλεύθηκε με το Κοινοβούλιο ο Πρόεδρος θέλει να υποβάλει την αλλαγή αυτή για την απόψινή ατζέντα η έκθεση της κυρίας Βαλέρο θα εξεταστεί ως τέταρτο σημείο για την απογευματινή συνεδρίαση μετά από την δήλωση για την 20η επέτειο της ε, Ειρηνευτικής ε, Συμφωνίας του Dayton. Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση θα εγκρίνουμε αυτή την αλλαγή. Και τώρα ερχόμαστε στις τρεις εκθέσεις που έχουμε του κυρίου Γκουαλτιέρη για την παράταση της θητείας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι.